Κάτω από όλα αυτά, τώρα παρακαλώ να τηρήσουμε τους λεπτούς υγεία. Ψηφίζουμε. Πρώτον, Μπουρούντι. Η περίπτωση του Μπόμπουρου Γκουρίγκα. Έχουμε κοινό ψήφισμα. Ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Έγκρινατε. Κύριε Πρέντα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ήθελα πριν την ψηφοφορία για τη Σαουδική Αραβία να πω ότι το ΕΛΚΑ δεν υπέγραψε το κοινό ψήφισμα, απλώς γιατί σε μία παράγραφο οι συντάκτες του κοινού αυτού ψηφίσματος Κάνουμε μια προσέγγιση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ισλαμικό κράτος. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στη συζήτηση, ασφαλώς και στο ψήφισμά μας ε, αντιτιθέμεθα σε κυρώσει κατά του Ραϊφ Μπανταουί. Ο μόνος λόγος ε, δηλαδή που δεν υπερψηφίζουμε το κοινό αυτό ψήφισμα είναι ότι οι συνάδελφοι έχουν κάνει αυτή την προσέγγιση Σαουδική Αραβία με Ισλαμικό κράτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το σημειώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι σε δική Αραβία που είναι η περίπτωση του Ραϊφ Μπαταουί. Κοινό ψήφισμα λοιπόν από έξι πολιτικές ομάδες. Πέντε, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της οφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στο H, ήταν στο αρχικό κείμενο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. M. Τώρα στο αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επόμενο για τα δέλτα δηλαδή είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε και περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Είναι η ομαδική τάφη των αγνώμενων της Άσιας. Υπάρχει κοινό ψήφισμα από 7 πολιτικές ομάδες. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Η τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί, οπότε ψηφίζουμε ολόκληρο το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Εκ μέρους των 191 που συνυπέγραψαν την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή όσον αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις, θέλω να επιστήσω σε ένα διαδικαστικό την προσοχή σας, παρακαλώ. Ο πρόεδρος του Σώματος αποφάσισε από μόνος του να μην ψηφίσουμε την πρόταση 191 συνυπογραφόντων εδώ, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι ο κανονισμός προβλέπει ότι ο Πρόεδρος πρέπει να υποβάλει σε ψηφοφορία στο σώμα με θετική ή αρνητική σύσταση, όπως θέλει, την αρχική πρόταση. Δεν έγινε όμως αυτό. Και πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και εμείς επιφυλασσόμεθα να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. După o decizie. Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι μία απόφαση που πήρε η διάσκεψη των Πρόεδρων και είναι το μόνο σώμα που μπορεί να αποφασίζει για αυτά τα ζητήματα. Και έτσι προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία. Προπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2. Διανατάσεως της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε για την απόφαση στο σύνολό τη. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στο θέμα ορισμών στην ειδική αυτή επιτροπή. Δεν έχω λάβει κάποιες ε, τροπολογίες για τους ε, διορισμούς στην επιτροπή αυτή. Οπότε δεν θα γίνει ψηφοφορία. Περνάμε. Κρίνεται χωρίς ψηφοφορία. Τώρα περνάμε στην ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα από έξι πολιτικές ομάδες. Τροπολογία 4. Διανοτάσεως χειρός παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 στο αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Δεύτερο μέρος, διανατάσεως της χειρός υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τροπολογία 5 διανατάσεις χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία σας. Εγκρίνεται. 20. Διανατάσεως χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23 από το αρχικό κείμενο μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 διανατάσεις της χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 δυνατά ισχυρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εκτιμώντας κάπα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή Τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα υπέρ, κατά, αποχές, νεκτή. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Îi rog pe colegi, îi rog pe colegi să ne lase să continuăm ședința. Συνάδελφοι, παρακαλώ να φύγετε ησύχω για να μπορέσει να συνεχιστεί η ολομέλεια. Domnul Arnet are o, un punct de ordine. Ο κύριος ε, Ανέτα ναι, έχει το λόγο για διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα προφορικώς να κάνω μια εξήγηση ψήφου για την περίπτωση του Ραΐφ Μπαντάουι. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας για την αντιπροσωπεία μας δεν θα είχαμε υπερψηφίσει αυτό το ψήφισμα, αλλά σε αυτή την περίπτωση υπερψηφίσαμε διότι η ανθρωπιστική διάσταση ήταν τόσο κατεπίγουσα. Πάντως, εάν δεν μπορούμε να έχουμε προφορική εξήγηση ψήφου, είναι σαν να αρνόμαστε, αρνούμεθα να πούμε στους πολίτες ε, της Βρετανίας, να αρνούμεθα να τους εξηγήσουμε τι, γιατί πράξαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πρόεδρος, ε, μου λένε ότι δεν θα υπάρξουν εξηγήσεις ψήφου για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Για αυτό το ψήφισμα μάλλον. Ε, δεν μπορούμε να περάσουμε σε εξηγήσει ψήφου για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Τώρα εγκρίνουμε τα διαδικαστικά, το, ε, συγγνώμη, τα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης. Εάν δεν έχετε